Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like... Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της κοινή συνεδρίασης των Επιτροπών μας ΑΦΕΤ ανάπτυξη και προϋπολογισμού σημείο 1, έγκριση της ημερίας διάταξης. Έχετε σχόλια. Μάλιστα. Ο κύριος Κασάλντο. Όχι. Για ποιο μετά. Ναι, ναι, ξέρω. Πάντα μιλάτε, το γνωρίζω σε όλα τα θέματα. Right, then we come to the chair's announcements. There of course none. We come to number three. Να περάσουμε στο σημείο 3. Έγκριση πρακτικών. Όχι. Εφόσον όχι, δεν ε, υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Έχουμε το ΕΤΒΑ. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. ΕΤΒΑ. Ε, λέμε για... Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο επενδύει στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στην ε, Αφρική. Τις τελευταίε ε, εβδομάδες οι επιτροπέ μας είχαν ανταλλαγές απόψεων με την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Εξωτερική δράση ε, και παρουσίασαν τα σχέδια έκθεσής του. Έχουμε τώρα 386 νομοθετικές τροπολογίες που πρέπει να εξετάσουμε εν ώψη τη ψηφοφορία που είναι προσχεδιασμένη για τις 24 Απριλίου. Πριν να ζητήσω από του να παρουσιάσουν την εργασία του θα στραφώ στου συμπροέδρου, τον κύριο Αρτουή και στον κύριο Πόγκα. Μηπω θέλετε ως πρόεδρε να προσθέσετε δύο λόγια. Κύριε Αρτουή δεν θέλετε. Μωρή, ούτε. Ωραία. Okay. Please, go ahead. Ε, ναι, παρακαλώ. Ε, χωρίς μικρόφωνο ο κύριο Αρτουή. Δεν ακούγεται. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Αρτουή, μάλλον δεν λειτουργεί αυτό το μικρόφωνο. τώρα λειτουργεί. Σας ευχαριστώ που μα υποδέχεστε για αυτή τη τέταρτη κοινή συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Θα ήθελα να χαιρετήσω τι προσπάθειε των εισηγητών και των σκιωδών. Λειτουργεί τώρα το μικρόφωνο. Μάλιστα λειτουργεί. που επεξεργάστηκαν ε, τροπολογίες και προετοιμάζουν και συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Να θυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε επικοδομητικό πνεύμα και πνεύμα ενότητος, διότι Χρειαζόμαστε ένα κοινοβούλιο ενωμένο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Δεν έχω όμω καμία αμφιβολία ότι θα επιτύχουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στους τρεις συνεισηγητές, κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ, Κούκαν και Φρουτζουλίτσα. Ποιο θέλει να πάει πρώτο στο λόγο, εσείς συμφωνήσει κάτι μεταξύ σας? Όχι, τότε οι κυρίες προηγούνται. Η κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις προέδρους και όπως ήδη ακούστηκε έχουμε ακόμα μια φορά συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Θα είναι μάλιστα η τελευταία συνεδρίαση που θα κάνουμε πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία μετά από την Πράσινη Εβδομάδα και γι' αυτό θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές γιατί κάναμε περίπλοκη εργασία, καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ωράρια και μετά για ιδέες και τρίτον ε, για το πώς να συντάξουμε όλε αυτέ τι ιδέες και να τι παρουσιάσουμε, αλλά πιστεύω πώ τα καταφέραμε. Ήταν λιγότερο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Έχουμε ήδη εμπειρίε ε, για το πώ λειτουργούν οι κοινέ επιτρο... επιτροπές και με τρει κοινές, ε, μάλλον επιτροπές ήταν ακόμη πιο δύσκολο, αλλά τελικά καταφέραμε μέσα σε αυτό το πνεύμα συνεργασία και ενότητα που έλεγε και ο πρόεδρος Σαρτουή Και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω και του συναδέλφου συναδέλφου, Όπως είπατε, υπέβαλαν 386 τροπολογίες. Ήταν ε, ισχυώδης, πολύ, πολύ επικοδομητική στην επεξεργασία ε, συμβαστικών ε, και ελπίζω πως στις 24 θα φανεί πόσο επικοδομητικό ήταν το πνεύμα και, ο στόχος και ότι ο στόχο του Κοινοβουλίου δεν είναι άλλο από το να βελτιώσουμε το κείμενο που έχουμε στο υποσυζήτηση. Να ευχαριστήσω και τις ε, πολιτικές ομάδες και την Επιτροπή, τις ε, γραμματείες μάλλον των τριών επιτροπών, γιατί πρέπει να δουλέψουμε και μέσα στους νέους κανόνες ε, του Κοινοβουλίου. Στόχος ήταν να απλοποιήσουμε λοιπόν την εργασία μας και ε, γι' αυτό και χρειάστηκε να προσαρμοστούμε. Ήταν περίπλοκο από τη μια πλευρά γιατί ήταν πολλοί κόσμοι που έπρεπε να συμφωνήσει και πολλέ τροπολογίε, αλλά πιστεύω πω όλοι δουλέψαμε με το, μέσα στο ίδιο πνεύμα και με τον ίδιο στόχο. Και ότι έτσι τώρα έχουμε μπροστά μα μια καλή συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τελειοποιηθούν, αλλά πάντω το σκελετό του συμβιβασμού τον έχουμε ήδη και έχουμε 25 συμβιβαστικέ τροπολογίε, αυτέ που έχουμε υποβάλει στο όνομα των τριών συνεισφέρων εισηγητών και που βελτιώνουν το κείμενο. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες γιατί ήδη τα έχουμε συζητήσει αρκετέ φορές, αλλά μόνο να πω και να τονίσω ότι στις εμβαστικέ τροπολογίες αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε τον ορισμό της προσθετικότητα additionality, που ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά του κειμένου ε, και να διευκρινίσουμε τους τελικούς στόχους. Επίση, ε, ε, περισσότερο μιλήσαμε και ορίσαμε τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Καθορίσαμε καλύτερα τι πολιτικέ για το δύο φύλλα και επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, προσθέσαμε και πίνακα επιδόσεων ε, που το χρησιμοποιήσαμε και όταν δουλέψαμε για το Ταμείο Εύση είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε ένα είδος δικτών που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τα υποψήφια project αλλά και για να εξασφαλίσουμε ότι όντως πληρούνται τα κριτήρια τα οποία θελήσαμε να θεσπίσουμε με αυτόν τον κανονισμό. Επίσης, ε, δώσαμε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να υποβάλει η Κομισιόν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και έτσι θα μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση και τις λεπτομέρειες του Ταμείου και εδώ το συμπληρώσαμε το διατακτικό, το άρθρο 17 αν θυμάμαι καλά, που αφορούσε τη διαφάνεια και την ενημέρωση για το εισέλογο εκθέσεις. Να επαναλάβω δε άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου στους συνεισηγητές και τους κοιόδης για την εργασία τους. Ε, πρέπει να τελειοποιήσουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά είμαστε σχεδόν σε τελική φάση. Ε, ώστε μετά από το Πάσχα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε Προσπαθήσαμε να συνονιθούμε για να έχουμε κοινή σύσταση στον κατάλογο ψηφοφοριών ανάμεσα στους τρεις ε, συνεισήγητες. Ε, πάντως μπορώ να σας πω ότι μ, κοινή θέση έχουμε και ε, θα φτάσουμε και στη συμφωνία εκεί που υπάρχουν ακόμα κάτι ψηλοδιαφωνίες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ συνάδελφε, ο κύριος Κούκαν, ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ε, ε, ε, ισχυρό προεδρείο έχουμε σήμερα. Εγώ εκτιμώ τα όσα μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού που είπε ότι που μίλησε με πολύ θετικό και επικοδομητικό τόνο και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα θέματα στις μελλοντικέ μας διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η συνάδελφος Καρδία Δαμπάλ ε, ανέφερε πολλά πράγματα, γι' αυτό και εγώ θα είμαι σύντομος, δεν έχω πρόβλημα με τα όσα μας είπε. Ε, να εκφράσω την εκτίμησή μου επίσης για τη συνεργασία με τους συνεισηγητές γιατί είχαμε πολύ επαγγελματικές συζητήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση. Δύο σημεία εγώ θέλω να αγγίξω σε αυτές μου τις εισαγωγικές παρατηρήσεις ότι πρόκειται για την τέταρτη περίσταση όπου οι τρεις μας επιτροπές ΔΕΒΕ, Budget και ΑΦΕΤ συζητάμε αυτό το θέμα από κοινού. Είναι δύσκολος και απαιτητικός ε, φάκελος όχι μόνο από την άποψη της διαχείρισης του αλλά και ως προς το περιεχόμενο του Στην αρχή θα, θα ήθελα να επαναλάβω εν συντομία κάτι που έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη θα έπρεπε να είναι ένα καινοτόμο ε, χρηματικό το πιστοτικό μέσο και θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, στις στοχές χώρες. Με το ΕΤΒΑ θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Αλλά αυτό το μέσο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως, μόνο ως αναπτυξιακό μέσο, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το μέσο ε, βασίζεται στις εγγυήσεις προς ιδιώτες επενδυτές και ότι χρειάζεται να προσελκύσουμε κεφάλαιο στις ε, χώρες αυτές και σε τομείς όπου υπάρχει ψηλός κίνδυνος και όπου διαφορετικά δεν θα γίνονταν επενδύσεις δηλαδή. Νομίζω πως έτσι ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, να μιλάμε ε, για την ιδέα της της ομαλής διαχείρισης αυτού του μέσου. Είπαμε ότι είχαμε πολλές τροπολογίες. μέχρι στιγμής... Ε, έχουμε, δουλέψει για κάποιες τροπολογίες. Ε, ε, είναι σημαντικό να εξισορροπήσουμε το, την, τη στοχοθέτηση και να δουλέψουμε αποτελεσματικά Ε, να είμαστε σαφείς ε, στους στόχους μας, όχι να υπερφορτώσουμε με επιπλέον στόχους. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ με τη διεύρυνση ε, αυτών των στόχων αυτών του μέσου. Να υπάρξει διάκριση ανάμεσα αυτού του μέσου και της αναπτυξιακής βοήθειας εν γέννη. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το μέσο είναι συμπληρωματικό στα άλλα αναπτυξιακά μέσα, και θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετική λογική. Είναι σημαντικό να προβλέψουμε αποτελεσματική εγκατάσταση αυτού του μέσου, πράγμα που θα σημάνει ε, αποτελεσματική δυνατότητα διακυβέρνησης χωρίς ε, περιτά, περιτό φόρτο, να μην δημιουργηθούν περιπλέον ε, φραγμοί ε, ούτε να είμαστε πολύ περιοριστικοί ε, χωρίς ε, να είμαστε περιοριστικοί λοιπόν για το δημόσια όργανα αλλά με το στόχο να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση ειδικά για τα μικρές και μεσές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλω να έχουμε σωστό κοινοβουλευτικό έλεγχο και γνώση για τις αποφάσεις που αφορούν ε, τις στρατηγικές που διέπουν αυτά τα μέσα. Ε, αυτές είναι οι αρχές λοιπόν τις οποίες έχω ακολουθήσει όταν ε, συζητήσαμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και όταν συζητήσαμε επίσης για τις υποδείξεις στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν εδώ συνεργαστήκαμε, είχαμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα μέσο το οποίο <coughs> θα ανταποκριθεί στο ρόλο για τον οποίο φτιάχτηκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έντουαρτ Κούκεν. Ο κύριος Φρουτζουλίτσα τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους άλλους δύο συνεισηγητές και όλους τους κοιόδες συζητητές για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Έτσι καταλήξαμε στις 25 συμβαστικές τροπολογίες. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα για το μέσο αυτό, κυρίως για την Αφρική και την Ανατολική Ευρώπη, για τις χώρες δηλαδή της ε, Ανατολικής Γειτονίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο πακέτο το οποίο θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης με οικονομική ανάπτυξη όπου θα συμμετέχουν όλοι, αντοχή κοινωνική και οικονομική των χώρων εταίρων. Θα στηρίξουμε επενδύσει και θα βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, συνεισφέροντα συγχρόνω στην εφαρμογή τη συμφωνία των Παρισίων και περιορίζοντα την μετανάστευση. Όσο προχωρούμε στην νομοθετική διαδικασία, θέλω να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που αναφέρονται και στην έκθεση, Πρώτα απ' όλα το στοιχείο της προσθετικότητας που διασφαλίζει ότι η ΕΤΒΑ θα συμφέρει σε δραστηριότητες οι οποίες αλλιώς δεν θα είχαν γίνει ή δεν θα είχαν μπορέσει να επιτευχθεί αποτελεσματικά στον ίδιο βαθμό χωρίς την στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με αυτός είναι και ο κύριος στόχος του ΕΤΒΑ. Υπάρχει και συμπληρωματικότητα όμως και η συνοχή που πρέπει να διασφαλιστούν στο σχέδιο αυτό εξωτερικών εγγύσεων βάσει των στόχων του 2030. Είναι σημαντικό το να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες που είναι ευάλωτες ή αντιμετωπίζουν συγκρούσεις. Χώρες που είναι ιδιαίτερα φτωχές. Λεβάνοντας υπόψη δηλαδή και το γενικό περιβάλλον και τις ικανότητές τους. Είναι πολύ σημαντικό ώστε να κρυθεί τελικά θεμητό το και θετικό το μέσο αυτό. Τα οικονομικά μέσα στο τοπικό νόμισμα ε, διασφαλίζουν την αποφυγή των διακυμάνσεων. Πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο που θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δράσεων του, των εκείσων ΕΤΒΑ και του Ταμείου εκείσων ΕΤΒΑ. Τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσφέρουν πληροφορίες και για επενδυτικές δυνατότητες του ΕΤΒΑ όταν επικοινωνούμε την κοινωνία των πολιτών με τον επιχειρηματικό κλάδο και γενικότερα τις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στο σημαντικό αυτό σχέδιο και πάνω απ' όλα τους άλλους συνεισηγητές, τους σκιώδες εισηγητές, τους επιρογνώμονες και τους βοηθούς μας. Τέλος, καλό Πάσχα σε όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ακούσαμε τους τρεις εισηγητές. Τώρα, έχω ζητήσει το λόγο. Επτά συνάδελφοι και σκιώδης εισηγητές. Θα διαβάσω τα ονόματα, μήπως έχουμε ξεχάσει κάποιον. Right. The names are Mr. Ponga, Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Kermel, Ms. Yetinemäki, Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12.30. 12.30 πρέπει να τελειώσουμε, έτσι. Κλείνει ο κατάλογος ομιλητών και σας παρακαλώ το πολύ δύο λεπτό καθένας, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ο κύριος Πόγκα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θέλω να πω, όπως είπαν και άλλοι πριν από μένα, ότι υπογραμμίζω το καλό έργο που επιτέχθη σχετικά με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές, τους χιώδες εισηγητές για τις συμβαστικές λύσεις τις οποίες καταλήξαμε. Μία παρατήρηση έχω να κάνω για την τροπολογία 313 που υπέβαλα με άλλους ευρωβουλευτές από την ΤΕΒΕ και που λέει ότι όταν είναι δυνατόν πρέπει το έτβα να μπαίνει κάτω από μια άλλη επιλεγμένη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση η τροπολογία εκεί, για γιατί πιστεύω ότι έτσι διασφαλίζεται η προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνοχή των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Πόστ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αρχίζω με ευχαριστίες προς τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, που ήταν όλοι ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις εκθέσεις που συμμετέχουν σε μία νομοθετική έκθεση. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ κάποια σημαντικά στοιχεία πάνω από όλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΕΤΒΑ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναφέρει το άρθρο 21. Αυτό συνεισφέρει επίσης και στις πολιτικές, στις αναπτυξιακές και γειτονίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απάλληψη της φτώχειας, την εξοπλική εργασία, τις ίσες ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει δηλαδή τις κύριες ρίζες της μετανάστευσης και να ενισχύσει το κράτος δικαίου την ε, χρηστή διακυβέρνηση και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας επίσης την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της πρέπει να αποτελέσει επίσης προτεραιότητα στα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΤΦΑ. Χρειάζεται παραδειγματική διαφάνεια επίσης σχετικά με τις πληροφορίες προς τους δικαιούχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει και το ίδιο υποκαθεστώς παρατηρητή και ο παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις. είναι ζωτική σημασία. Επίσης, το μέσο αυτό να είναι συμπληρωματικό με άλλες πρωτοβουλίες. Και βέβαια υπάρχει διάκριση ανάμεσα στι δραστηριότητε αυτές και εκείνες τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, γιατί οι συνάδελφοι έφεσαν τα άλλα ζητήματα. Θα επικεντρωθώ στην ανάπτυξη και τι εξωτερικέ υποθέσει. Εμεί από την ECR θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πηγή της μετανάστευσης. Νομίζουμε ότι αυτό το θέμα είναι βασικό σημαντικό καινούριο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να αποσυντονιζόμαστε από το στόχο μας. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο πώς αντιμετωπίζουμε τις βασικές αιτίες. Αν βάλουμε πολλές ε, πτυχές θα χάσουμε από το προσκήνιο αυτά που πρέπει πραγματικά να γίνουν. Όπως είπαν και οι συνεισηγητές, είναι πολύ σημαντικό ε, να μην έχουμε πολλές εναλλακτικέ ε, θεωρήσεις και να προσπαθήσουμε να δούμε όλα τα καλά που μπορούμε να κάνουμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να έχουμε κάτι το οποίο δεν θα επιτύχει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε και καλή αξιολόγηση του μηχανισμού για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια καταπανώνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ότι αποφεύγονται τα λάθη του παρελθόντος και για να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Γέτεν Μέκη, τώρα εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που ο Πρόεδρος κύριος Αρτουή έχει θεωρήσει ότι πρέπει να ε, στοχεύσουμε σε μια κοινή συνεργασία η οποία είναι εξαιρετική αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι ένας από τους ε, λόγους, τους πιο διαδεδομένους ε, που οδηγούν στη μετανάστευση. Νομίζω ότι στο μέλλον η κλιματική αλλαγή θα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν θεσπίσει στόχους που είναι πολύ ε, μη φιλόδοξοι, πολύ χαμηλοί. Θα μπορούσαμε να τους αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι πιο φιλόδοξο. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχει να κάνει με αυτά που συνέβησαν μεταξύ 2006 και 2012, την τεράστια ξηρασία που οδήγησε σε τεράστια μεταναστευτικά κύματα. Φυσικά δεν είναι η ξηρασία που προκάλεσε μόνο τη μετανάστευση, αλλά είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς λόγους. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μεγάλη ποσότητα αυτών των κονδυλίων για να χρηματοδοτήσουμε μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος του FC είναι 40% και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει στόχο 50%. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ λοιπόν ότι το καθιερωμένο επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αυξηθεί. Αυτά είχα να πω. Thank you, dear colleague. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Η κυρία Χάουταλα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Συμπρόεδρε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ δρόμο και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυξιακές προσπάθειες η δουλειά που έχει γίνει ως τώρα ε, είναι μια δουλειά που ικανοποιεί την ομάδα μου σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω όταν μιλάμε για την ψηφοφορία στις 24, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την προσθε... προστιθέμενη αξία, την προσθετικότητα και συμπληρωματικότητα αυτού του εργαλείου, γιατί δεν πρέπει να δαπανίσουμε και να σπαταλίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων χωρίς να υπάρχει ένα εργαλείο εγγύσεων. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά κάποιες ψηφοφορίες, κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως ε, να μην θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Ε, τα ορυκτά καύσιμα, κάποια φράγματα, υδροηλεκτρικά. Αυτά είναι πράγματα ε, που δεν θα θέλαμε να χρηματοδοτήσουμε με ένα εργαλείο που έχει θεσπιστεί για να πατάξουμε τη φτώχεια φτώχεια. Επίσης, ε, υπάρχει η τροπολογία 54 των Πρασίνων ε, για την, το μηχανισμό παραπώνων, για να μπορούν να προσφύγουν όσοι έχουν πληγεί από ένα project. Επίσης, αν υπάρχει οποιαδήποτε αίσθηση καθή, ε, επίγοντος, θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα γιατί πραγματικά κανένας άλλος δεν θα είναι τόσο φιλόδοξος όσο εμείς. Ευχαριστούμε τη Χάλντι Χάουταλα και ο κύριος Καστάλντο για το FDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την θέση που έχουμε για αυτήν τη σημαντική κοινή έκθεση την οποία βεβαίω χαιρετίζουμε θετικά και με αισιοδοξία. Ε, το ΕΤΒΑ και η εγγύησή του θα πρέπει να είναι ο πρώτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικές επενδύσεις, ένας πυλώνας με μιας ε, μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των, ε, για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων και για να κατανοήσουμε τα αίτια της μετανάστευσης. Θα πρέπει να έχουμε ωστόσο κάποιες μήνυμου προϋποθέσεις, ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είμαστε κατά των ιδιωτικών επενδύσεων βεβαίως, αλλά θέλουμε δεν θέλουμε να ε, ε, ηγηθούν του παιχνιδιού οι πολυεθνικές, αλλά ε, να μπορέσουν να ωφεληθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, να μην εστιαστούμε μόνο σε μεγάλα έργα υποδομής που έχουν ε, έχουν αυτά βέβαια μεγάλο αντίκτυπο στην απασχόληση, αλλά να μην είναι επίμαχα από καμία άποψη, ούτε την περιβαλλοντική, ούτε την οικονομική, ούτε την κοινωνική. Και θέλουμε μια ανεξάρτητη εξάντε εκτίμηση για το κόστο και την ωφέλεια. Επίσης, ε, λογοδοσία πλήρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα και στου Ευρωπαίου πολίτε, δίνοντα ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των τοπικών ε, κοινοτήτων. Οι πληθυσμοί εξάλλου είναι αυτοί, οι εντόπιοι πληθυσμοί είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση και πάντοτε θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση μαζί τους στον καθορισμό των project αυτό ισχύει και για την χορήγηση των χρηματοδοτήσεων. Ο στόχο θα είναι να ανεπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα ο τοπικό, γιατί χωρί αυτή την ανάπτυξη ποτέ δεν θα δημιουργηθούν οι απαραίτητε προποθέσει για την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη που μακροπρόθεσμα θα μπορέσουν να αναχαιτήσουν τη μετανάστευση. Δεν θα πρέπει πάντω να είναι πέρασμα χρημάτων προ ε, του φορολογικού παραδείσου. Η έκθεση τη ΕΤΕΠ δείχνει πω αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτές είναι οι μήνυμοι απαιτήσει που θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν, γιατί διαφορετικά θα είναι μια νιωστή αποτυχία της πολιτικής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Τελευταίοι δύο ομιλητές. Κέγγε πρώτα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ξεκινώ ευχαριστώντας ε, τους ε, συνεισηγητές που εργάστηκαν εντατικά για το πρόγραμμα αυτό και για τη δημιουργία αυτού του ταμείου. Γιατί αυτό το ταμείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τελικά ε, στόχο έχει για να, μπορέσουμε να επενδύσουμε ε, ώστε να εκριζωθούν τα βαθιά τεραέτια που πλήττουν πολύ κόσμο και αναγκάζουν τον κόσμο να φεύγει από τη χώρα του. Ε, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση αλλά και στα project για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό το Ταμείο θα δώσει την ευκαιρία να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη για όλους, αλλά και να είναι και βιώσιμη σε πολλούς τομείς. Μία από, τα, ένα από, τα, από τις πληγές Αφρικής είναι η ανεργία των νέων και η δυνατότητα να μπορούμε να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για νέους και παιδιά είναι πολύ σημαντική και να προσπαθήσουμε επίσης να εγγυηθούμε δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Αλλά για πρώτη φορά βλέπω και άλλη μια σημαντική πτυχή, τη ψυχή της ε, αντοχής και της διατροφικής ασφάλειας. Ε, τέλος, ε, κάτι που μας αφορά εμάς κυρίως και αφορά την συμβιβαστική της 25, ρόλος του Κυπροκοινοβουλίου, έχοντας υπόψη ότι υπάρχει και η ΑΚΕ, η ισομερή Συνέλευση ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το ταμείο. Να μην περιοριστούμε δηλαδή μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό το βλέπω πολύ θετικά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά το κοτονό ενισχύοντας την, ε, τον ρόλο της Ισομερού Συνέλευσης ΑΚΕ Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Κέρνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον, ε, τους συνεισηγητές για τη δουλειά τους. Νομίζω ότι για όλα όσα υπόθηκαν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αυτή η έκθεση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ειδικά στην Αφρική για να προλάβουμε την τα ρεύματα της μετανάστευσης και θα πρέπει να έχουμε το θάρρος όχι μόνο να φύγουμε το θέμα, αλλά να βρούμε μια ε, και να απαιτήσουμε μια λύση για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει κάποια βασική ιδέα για αυτό το θέμα, μια έννοια. Αυτό μπορεί να είναι ένα λιθαράκι, αλλά δεν υπάρχει το, η γενικότερη έννοια. Τώρα, πέρα από αυτά, εγώ αμφισβητώ τη δυνατότητα χρηματοδότησης εγγυήσεων και κατά πόσο ε, φτά, μπορεί αυτές να φτάσουν μέσα από ένα σύστημα τραπεζικό για να πετύχουν αυτό που θέλουμε. Μιλάμε για περισσότερη ε, διαφάνεια, όμως ταυτόχρονα έχουμε εδώ ένα σύστημα χρηματοδότησης το οποίο δεν μας δίνει καμία διαφάνεια. Εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για την προσθετικότητα και θέλουμε το ένα να το συμπεριλάβουμε και το άλλο να το εξαιρέσουμε. Όμως όλα αυτά ε, δεν ε, τα έχουμε καταφέρει. Εμείς πρέπει να επενδύσουμε στην, στην Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε μετά να δούμε ακριβώς πώς θέλουμε να προχωρήσουμε μέσα από άμεσες επενδύσεις προς την εκπαίδευση και τις υποδομές. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Αυτή ήταν η λίστα με όλους τους συναδέλφους που θέλησαν να μιλήσουν. Τώρα ζητώ από τους εκπροσώπους της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων να μας πούν εάν θέλουν να τοποθετηθούν. Μπορείτε να μας δώσετε το όνομά σας και τη θέση σας. Γεια σας, είμαι υπεύθυνο ε, στην DG DEFCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, καταρχάς, να ευχαριστήσω τις τρεις επιτροπές για την εξαιρετική εργασία τους ε, και για τον ε, μεγάλο αριθμό, αλλά ιδιαίτερα επικοδομητικό των τροπολογιών υπάρχουν πολλές τροπολογίες σχετικά με την προσθετικότητα. Μπορεί τα στάνταρ να είναι τα υψηλότερα που έχουν ποτέ ε, τεθεί σε οποιοδήποτε ε, εργαλείο ανάπτυξης και συνεργασίας. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες. Επίσης υπάρχει η ανάγκη για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχουν ίσως κάποια μόνο κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τη δική μας άποψη κάποια θεσμικά που έχουν να κάνουν με την ε, ε, εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στο Επιχειρησιακό Συμβούλιο, ας πούμε, και ένα που έχει να κάνει με τα, με τα σκέλη επενδύσεων και τις ε, πράξεις εξουσιοδότηση. Αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή, αλλά όμως θέλουμε να έχουμε ανδρωθεί και για τις θεσμικές σειράξεις. Είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή, ελπίζω και φαντάζομαι και για την EIS, να δώσει τα πρώτα από τα αποτελέσματα τον Νοέμβρη στην ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, για να δείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει γρήγορα όταν χρειάζεται. Είναι δύσκολο το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας. Τα πρώτα ε, σκέλη επενδύσεων μετά από συναντήσεις του Στρατηγικού και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ε, είναι ε, τα πρώτα που θα ε, δοθούν. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε αυτά τα θεσμικά όργανα ως πρεσβευτές που θα προωθήσουν αυτό το project εγκαίρως για την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής το Νοέμβρη. Έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, η το χρονοδιάγραμμα για την τριμερή διάσκεψη μπορεί να μην μας επιτρέψει να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε πριν το καλοκαίρι. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τους συναδέλφους από την νομική υπηρεσία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο διαδικασιών, γιατί το timing είναι πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό να γίνει πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και αν μπορεί κάποιος εδώ να συνεισφέρει σε αυτό, για να πετύχουμε αυτό το στόχο, όλοι θα βοηθούσε. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχετε κι εσείς να πείτε κάτι, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Φραντσέσκα Ρεμόντι ονομάζομαι και εκπροσωπώ εδώ τα συνολικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όπως καταλαβαίνετε, τα κύρια μηνύματα τα μετέφερε ήδη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για μας είναι σημαντικό το χρονοδιάγραμμα. Για να αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά και με τους δικαιούχους, με τις χώρες εταίρους. Είναι και για αυτούς πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στις αποφάσεις. Όπως ξέρετε, οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το Στρατηγικό Συμβούλιο ελπίζουμε ότι θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις διαβουλεύσεις μαζί τους. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Οι συνεισηγητέ θέλουν να πούνε κάτι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώ τότε σα υπενθυμίζω ότι θα ψηφίσουμε τη Δευτέρα 24 Απριλίου στι 5.30. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρόεδρε, Μωρή, παρακαλώ. Όχι. Εντάξει, έληξε λοιπόν η συνεδρίαση και μάλιστα 10 λεπτά νωρίτερα. Καλό μεσημέρι.